έχουμε μια σύντομη σύγκριση της εκθέση Και η όσον αφορά την ε, προβληματική, τη θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία ναι. Επίτροπε, μέχρι τώρα η γενική και επαγγελματική αεροπορία δεν αντιμετωπιζόταν σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Βλέπουμε όμως να υπάρχει μια ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής ε, της γενικής και εμπορικής αεροπορίας και γίνεται ένας και πιο, όλο και πιο σημαντικός ε, κλάδος. Έχουμε ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, ο αριθμός ε, των ε, σκαφών διπλασιάστηκε από το... 2005 και από το 2006 και ε, πάρα πολλές θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τον τομέα αυτό. Με την γενική αεροπορία ε, τα τελευταία 10 χρόνια θα έχουμε 30 με 50 χιλιάδες ε, σκάφη που θα καταχωρηθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο της αεροπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτονται διαφόρων ειδών ε, μεταφορές που έχουν ε, ε, οικονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον, ευέλικτες μορφές μεταφοράς, παραδείγματος χάρη, έχει να κάνει επίσης με τις θύσεις για αναψυχή, με την ιδιωτική μεταφορά, μεταφορά για επαγγελματικού σκοπούς. Αναπτύσσονται επίσης ικανότητες αεροπορικές που αξιοποιούνται μετά στην αεροπορία γενικότερα. Αυξάνεται όλο και περισσότερο ο τομέας αυτός ε, και ε, ο αντίστοιχο λοιπόν τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 16% τη παγκόσμια αγορά και αξίζει κάποια υποστήριξη. Ε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συλλέξει στοιχεία, να συλλέξει δεδομένα ε, τα οποία θα δοθούν σε αυτούς που θα λάβουν τις αποφάσεις. Χρειάζονται οι κατάλληλες στατιστικές πληροφορίες ώστε να ληφθούν σωστές αποφάσεις για την γενική και εμπορική αεροπορία. Δεύτερον, ε, πρέπει να ε, σεβαστούμε την αρχή της αναλογικότητας σε οποιασδήποτε νέες ρυθμίσεις και κανονισμούς που θα ε, προκύψουν. Οποιοδήποτε, τέτοιοι κανονισμοί θα πρέπει να είναι ε, κατάλληλοι για τα πολύ μικρά μονοθέσια αεροσκάφη. Ε, και το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν πρότυπα και κανονισμούς που θα ισχύσουν. Βεβαίως ταυτόχρονα θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν εις βάρος της ασφάλειας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι κανόνες της ε, ε, αξιοπλοίας που ε, έχουν ήδη υιοθετηθεί ότι δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν, να αποδυναμωθούν. Τρίτο σημείο, η πρόσβαση στον ενέργειο χώρο και στα μεγάλα ε, αεροδρόμια για την ε, γενική και εμπορική αεροπορία, ιδιαίτερα ε, στο περιφερειακό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν η γενική και εμπορική αεροπορία να έχει την απαραίτητη πρόσβαση και να έχει και τα κατάλληλα σλότ, τις χρονοθυρίδες προς απογείωσης. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί έτσι ο κλάδος αυτός θα εξασφαλίσει καλύτερη διασυνδέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Όσον αφορά το ΣΥΖΑΡ και τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, και εδώ πάλι θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε σωστούς και αναλογικούς ε, κανόνες που να αντιστοιχούν στα μικρά αυτά αεροσκάφη ε, της ε, γενικής και εμπορικής αεροπορίας. Τέταρτον, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τα μικρά αεροσκάφη βεβαίως παράγουν λιγότερη, μικρότερη ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα από ό,τι τα μεγάλα αεροσκάφη. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στα πλαίσια του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και της επιχείρησης Caesar. θα πρέπει να φροντίσουμε τα, όλα τα αεροσκάφη αεροσκάφη βεβαίω να είναι ε, λιγότερο, ε, να ρηπαίνουν λιγότερο στο μέλλον για να χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα. Η έκθεση αυτή ε, πιστεύουμε ότι ε, ε, οδηγεί σε ένα πραγματικά πλαίσιο, κατάλληλο πλαίσιο για την μελλοντική νομοθεσία για τον τομέα αυτό και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα εκφραστούν αύριο με μια συντριπτική πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία. Η κυρία Επίτροπος έχει το λόγο. And... Η Επιτροπή ευχαριστεί την εισηγητή και την αρμόδια κοινοβουλική αστυνομία για τη θαυμάσια εργασία. Τον ε, ε, Γενάρη 2008 στην Προετοίμασε η Κομισιόν μια εκθέση για το θέμα αυτό που συνοδεύτηκε από τα πρώτα συμπεράσματα του 2008 τον Απρίλιο και έχουμε τώρα την έκθεση αυτή του Κοινοβουλίου. Ο τομέα αυτό τη Γενική και Επανομική Αεροπορία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη και ε, βασίζεται επίσης σε πάρα πολύ έρευνα και ανάπτυξη και ναυτίσεται γιατί το 2 τρίτα των αεροσκαφών που είναι εγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εμπίπτουν στον τομέα αυτό. Η Γενική και Παλαιτική Αεροπατορία αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα πολύ διαφοροποιημένο τομέα και θα πρέπει η διατάξη διακανονισμού να είναι καλά προσαρμοσμένες χωρίς να διακυβεύουν τη ασφάλεια και πιστεύουμε ότι όλα αυτά τηρούνται από το Κοινοβούλιο στη έκθεση του. Τρει τομεί είναι εκείνοι που θα πρέπει να διατηρήσουν την προσοχή Η ανάπτυξη κοινών προτύπων ασφάλεια για την γενική ε, αεροπορία. Η έναρξη τη αεροπορία αυτή στη νέα γενιά διαχείρισης των αεροπορικών μεταφορών και μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του τομέα θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ενιαίο τομέα ασφάλεια για την μη εμπορική αεροπορία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν δίνεται μόνο επαρκές επίπεδο ασφάλειας, αλλά χωρίς να επιβάλλεται ιδιαίτερο βάρος στους ιδιοκτήτες αυτών των ε, επιχειρήσεων. Επίση, θα πρέπει να αναπτύξουμε το σύστημα MTS για την Ευρώπη, γνωρίζοντα ότι ο ενέργειο χώρο είναι ένα κοινό αγαθό που θα πρέπει να είναι ανοιχτό στη χρήση του σε όλου του ενδιαφερόμενου. Ο ως ευρωπαϊκός αερο... χώρος και το ΣΕΖΑΡ θα πρέπει να επιτρέψουν την ε, ισότιμη πρόσβαση στον ενέργειο χώρο και στα αεροδρόμια. Τέλο, η γενική και επαγγελματική αεροπορία παρόλο τι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχει επιπτώσει στο περιβάλλον και όπως γενικά οι αεροπορικέ βιομηχανίε θα πρέπει και αυτοί να μειώσουν τι επιπτώσει. Εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της αναλογικότητα. Η Κομισιόν προβλέπει στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο βάσει των αρχών της έκθεσης και η Κομισιόν θα σας παρουσιάσει προσεχώς την πρόοδο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ρέντινγκ. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία από τη έκθεση αυτή. Και περνάμε τώρα στην μια σύντομη παρουσία τη έκθεση Άννα Ζαμπορσκά για την ομαλυψία με βάση το φύλλο και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι,